Die Präsidentin! Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die Sitzung. Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Πρώτα θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι ο κύριος Γιώργος Παπακοσταντίνου και από σήμερα, 7η Οκτωβρίου, διορίστηκε υπουργό στην ελληνική κυβέρνηση. Του εκφράζω τα συγχαρητήριά μου, σημειώνω τον διορισμό του και σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της νομοθεσίας περί αμέσων εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 του κανονισμού διαπιστώνω την απελευθέρωση της έδρας του από την 7η Οκτωβρίου 2009. Από τη διάσκεψη των Προέδρων Πολιτικών Ομάδων έλαβα πρόταση για τον διορισμό των μελών της έκτακτης ε, επιτροπής για ε,